Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στη συνεδρίασή μα σήμερα. Να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας, γιατί θα ξεκινήσω τη συνεδρίαση. Λοιπόν, σας καλωσορίζω, θα, θα σήμερα Λοιπόν, να δούμε το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Πρώτα απ' όλα, έγκρισή της. Συμφωνείτε να την εγκρίνουμε χωρίς τροποποίησης. Δεύτερον, οι 20 γλώσσες ε, του γλωσσικού μας ε, προφίλ είναι διαθέσιμες, ε, αλλά όχι τα μαλτέζικα. Δεν θα έχουμε μαλτέζικη καμπίνα σήμερα. Καλώς ήρθατε. Μια άλλη ανακοίνωση. Έχουμε την 25η επέτειο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης. Θα έχουμε ένα γεύμα γι' αυτό στις 21 Νοεμβρίου, κατά τη μεσημεριανή διακοπή. Και περνάμε στο 3. Ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους. Και θα μας κάνει ενημέρωση η κυρία Ράντκα Μαξοβά. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ενημερώσω για τον πρώτο και το δεύτερο τριμερή διάλογο για την οδηγία για την απόσπαση των οδηγών. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έγινε την 1η Οκτωβρίου. Ήταν κοινός τριμερής διάλογος και για τα τρία θέματα. Πολιτικά τα τρία θέματα είναι στενά συνδεδεμένα. Το Συμβούλιο και εμείς συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε συμφωνία όσο ταχύτερα γίνεται ή δυνατόν κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας. Επίσης, συμφωνήσαμε επί των μεθόδων εργασίας και βεβαίως με βάση την ε, βασική αρχή ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα. Επίσης, ε, συμφωνήσαμε και ένα χρονοδιάγραμμα τεχνικών συναντήσεων και τις ημερομηνίες των διαλόγων, των τριμερών διαλόγων 4 και 5 Νοεμβρίου που έγινε λοιπόν και στο Στρασβούργο 25-26 ε, Νοεμβρίου. Ο δεύτερος τριμερής διάλογος μετά τις τεχνικές συνεδριάσεις ε, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Και μετά τις τεχνικές συνεδριάσεις η Φινλανδική Προεδρία υπέβαλε συμβαστικέ προτάσει για θέματα επί του οποίου το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν παρόμοιου πολιτικού στόχου, αλλά έχουν διαφορέ επί των κειμένων και από πλευρά προσέγγιση. Και επιτύχαμε ε, σημαντικέ επιτυχίε ε, στα επόμενα θέματα. Πρώτα απ' όλα, έλεγχο για, ε, για το χρόνο εργασία των οδηγών. Για το θέμα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστούν διάφορα τεχνικά θέματα, αλλά ε, επί της ουσίας συμφωνούμε. Δεύτερον, συστήματα ενημέρωσης. ERRU και II. Συμφωνήσαμε με την κατεύθυνση των συμβιβασμών, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστεί πώς θα υπάρχει απευθείας πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα στοιχεία για την αξιολόγηση του κινδύνου. Κατόπιν υπήρξε μια ενδεχόμενη συμφωνία για την, ε, για την δήλωση απόσπασης, γιατί θα πρέπει να διευκρινίσουμε πώς θα εντοπίζονται οι οδηγοί για να μην υπάρχουν ε, παραχαράξεις στοιχείων. Επίσης, η αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, το αριθμή μητρώου κοινωνικής ασφάλισης είναι κάτι που θα συζητηθεί αργότερα στον τρίτο διάλογο. Θα ψάξουμε λοιπόν για τρόπο πώς να μπορούμε μέσω κάτι που να είναι κοινό σε όλους να εντοπίζουμε, να δούμε ποιοι είναι ο οδηγός. Οι τρίτες χώρες είναι ανοιχτές για να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ των δικών μας εταιρεών και των εταιρεών τρίτων χωρών. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και θα συνεχιστεί. Το Συμβούλιο επέβαλε συμβαστικές προτάσεις. Το Κοινοβούλιο θέλει να τις εξετάσει περαιτέρω. Συζητήσαμε τη δυνατότητα να υπάρξει κοινή προσέγγιση της Ένωσης. Ένα άλλο θέμα που εκκρεμεί είναι τα, μάλλον διάφορα θέματα είναι η ευφυή επιβολή του νόμου, η υποβολή εκθέσεων και η κατάρτιση. Θέλουμε το Συμβούλιο να είναι λίγο πιο φιλόδοξο και ζητήσαμε να μα στείλει έγγραφα τα οποία ε, τα λάβαμε σήμερα το πρωί. Έχουμε σημαντικά πολιτικά θέματα που θα συζητηθούν στον τριμερή διάλογο στις 26 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων, θα συζητήσουμε για τις ε, αποσπάσεις για ε, τους οδηγούς λεωφορείων και για την εντόπιση, τον εντοπισμό των οδηγών από τις τρίτες χώρες. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Μαξοβά. Έχετε ερωτήσεις? Ο κύριος Βίλεμσεν. Κυρίε Γιονγκέριους. Και η κυρία Σάιμπη. Άλλος. Παρακαλώ. Ο κύριος Βίλεμος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια που μας ενημέρωσε. Μια σύντομη ερώτηση. Ένα βασικό κλειδί για να αποφεύγονται οι καταχρήσεις των εξαιρέσεων από τους κανόνες για, ε, την, ε, για, τους, για τις εξαιρέσεις, ε, το lex specialis, είναι η ευφυής ταχογράφη. Έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το σεβασμό των δικαιωμάτων των οδηγών φορτηγών για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης. Δεν ξέρω όμως αν θα έχουμε έτοιμη τεχνολογία όταν θα πρέπει. Ορισμένοι λένε πως δεν θα είναι. Άλλοι λένε ότι σίγουρα θα είναι έτοιμη η τεχνολογία όταν θα μεταφερθεί αυτή η οδηγία στις εθνικές νομοθεσίες. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει η Γητριά αν έχουμε πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στους τριμερείς διαλόγους για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιονγκέριους, ευχαριστώ πολύ. θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα οδήγηση και ανάπαυσης ε, χωριστά έτσι δεν είναι. Δεν το έχουμε στην μέσα διάταξη. Τότε θα μιλήσω γι' αυτό αργότερα. Τώρα η ερώτηση στην εισηγήτρια είναι η εξής. Μια από τις προτάσεις του Κοινοβουλίου για να εφαρμόζεται ο νόμος ήταν ότι θα πρέπει να αναρτώνται τα αποσπάσματα από τις πληρωμές για να έχουμε όλοι έλεγχο για το εάν και κατά πόσον ε, έχουν πληρωθεί όπως ε, έπρεπε. Δεν ξέρω, το συζητήσατε αυτό, δεν είπατε τίποτα γι' αυτό. Γιατί βέβαια μπορεί κανείς να λάβει μέσω του ίντερνετ ε, μία απόδειξη της πληρωμής του. Αν τα έχουμε όλα αυτά στο ίντερνετ ε, θα είναι πολύ εύκολο να ε, εξετάσουμε κατά πόσον έχουν εφαρμοστεί οι κανόνες. Ευχαριστώ. Θα το συζητήσουμε το θέμα που αναφέρατε χωριστά. Είναι το επόμενο θέμα. Η κυρία Σέμπλη η κυρία Σομπλή. Καλημέρα σας. Είμαι η συγγήτρια της Γκουε για το θέμα αυτό, χρόνος ανάπαυσης και οδήγησης. Και ε, να αναφέρω τα τρία θέματα που θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικά για τις επόμενες συνεδριάσεις που θα κάνουμε στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Όπως είπε και ο συνάδελφος Νικολά Βίλουμσεν, ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν οι ευφυείς τάχογράφοι θεωρούμε ότι είναι πολύ ουσιώδες ε, να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα τάχιστα. Αν θέλουμε συνθήκε εργασίες των ε, φορτηγατζίδων να γίνονται σεβαστές. Κάτι άλλο που θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδες. Η περίοδος αναφορά, αναφοράς για το χρόνο ανάπαυσης των οδηγών φορτηγών. Θέλουμε να διατηρηθεί η τροπολογία 379 του Κοινοβουλίου που λέει ότι η περίοδος αναφοράς πρέπει να είναι δύο εβδομάδες και όχι τέσσερις όπως προτείνει το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Και τέλος, τρίτο θέμα. Είναι να μπουν και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, τα φορτηγάκια, γιατί τώρα συμπεριλαμβάνονται μόνο όσα είναι άνω των 3,5 τόνων. Οτιδήποτε όμως είναι διεθνείς μεταφορές σε τέτοια μικρά φορτηγάκια κάτω από 3,5 τόνους είναι χωρίς κανένα κανόνα. Γι' αυτό προτείνουμε να διατηρηθεί η τροπολογία 373 του Κοινοβουλίου που καθορίζει τι θα γίνει για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Λέει κυρία Μάξοβα, όσον αφορά τους ευφυείς ε, ταχογράφους, είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε στους τριμερείς διαλόγους, είναι θέμα πολιτικής φύσεως και μιλάμε και για τη δυνατότητα να αναβληθεί η ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας και ξέρουμε ότι ταχογράφοι δεύτερης γενιάς δεν λειτουργούν πλήρως ακόμα. Τώρα, αυτές οι πληρωμές, αυτό είναι κάτι που δεν συζητήσαμε μέχρι τώρα. Και το τρίτο ερώτημα αφορούσε τα ελαφρά εμπορικά οχήματα. Το συζητήσαμε αυτό, αλλά αποτελεί ακόμα εκκρεμότητα. Για ποιο λόγο, διότι η οδηγή των ελαφρών αυτών εμπορικών οχημάτων καμιά φορά παραβιάζουν κανόνες και δημιουργούν κινδύνους για άλλους οδηγούς και αυτό στην επόμενη συνεδρίασή μας θα το συζητήσουμε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Μπορούμε να συνεχίσουμε με την, τον κανονισμό 561, τροποποιητικό κανονισμό του έτους 2006 που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσει για μέγιστη μερίσιο, μέγιστο ημερήσιο εβδομαδιο χρόνο οδήγηση και ημερήσιο και εβδομαδιο χρόνο ανάπαυση. Ο κύριος Ράτκε είναι εισηγητής και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανιστή. Καταρχάς, Χαίρομαι που δεν πρέπει να αναφέρω όλο τον τίτλο του θέματος κάθε φορά, γιατί θα μου έπαιρνε πολύ χρόνο, αλλά χωρίς αστιάκια. Είχαμε έναν κοινό τριμερή διάλογο και άλλους δύο τριμερείς διαλόγους. Συζητήσαμε όλα τα θέματα του πακέτου κινητικότητας και έναν τριμερή διάλογο είχαμε πιο συγκεκριμένα για τον χρόνο οδήγησης και τον χρόνο ανάπαυσης. Τι συνέβη μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η τριμερείς διάλογοι ήταν τεχνικής φύσεως και τα καυτά ζητήματα θα προκύψουν στο Στρασβούργο. Και γι' αυτό έχουμε μια ανοιχτή συνεδρίαση. Ε, ποια είναι τα καυτά θέματα. Η εβδομαδιαίος, εβδομαδιαίος χρόνος ανάπαυσης για τους οδηγούς που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και αν μπορούμε να έχουμε δύο σύντομε περιόδους που ενώνονται. Είχαμε πολλές συζητήσεις στο Συμβούλιο για το θέμα των υποδομών των αυτοκινητοδρόμων, χώρου στάθμευσης με άλλα λόγια, τουαλέτες κλπ. Και αυτά είναι θέματα πολύ στενά συνδεδεμένα με την απαγόρευση του να διανυχτερεύει κανείς στην καμπίνα του οδηγού, να μένει στο φορτηγό οδηγός. Όταν συζητούσαμε το θέμα στο Κοινοβούλιο, ήταν πολύ σαφές ότι όσο αφορά την απαγόρευση του να κοιμάται οδηγός στην καμπίνα οδήγησης, δεν ήταν ζήτημα άνεσης, αλλά ήταν θέμα ασφαλείας που ετίθετο. Και νομίζω ότι δοθέντος ότι η πλειοψηφία έχει συμφωνήσει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, οι οδηγοί να κοιμούνται και να διανυχτερεύουν σε αφύλακτους χώρους που δεν φωτίζονται, σε χώρους τάθμευσης ε, με αγαθά υψηλής αξίας. Αν αυτό αποφασίζει η πλειοψηφία, τότε τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν τις κατάλληλες υποδομές. Και όσον αφορά την επιστροφή τους, ήταν σαφής ο χρόνος αναφοράς και για τους εφίσταχογράφους ταχογράφους επίσης συζητήσαμε. Ίσως να μην προχωρήσαμε πάρα πολύ, αλλά εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είμαστε υπεύθυνοι για τεχνολογικές εξελίξεις. Τεχνολογικές εξελίξεις δεν έχουν προχωρήσει πολύ, αλλά εμεί είμαστε υπεύθυνοι για την νομοθεσία. Καμιά φορά πρέπει κανείς να νομοθετεί ούτω ώστε να ασκήσει κάποιες πιέσεις στις Τεχνολογίες εξελίξει απ' έξω. Και η επέκταση τώρα του πεδίου εφαρμογής για τα ελαφρά εμπορικά οχήματα μέχρι 2,5 τόνους, αυτό είναι σημαντικό να γίνει και να μην χάσουμε και τα πάντα, θα πρέπει να εστιαστούμε επί εκείνων οι οποίοι είναι επαγγελματίες ε, οδηγοί όπου η οδήγηση είναι στο επίκεντρο της δουλειάς τους. Να μην αρχίζουμε να ελέγχουμε και να τιμωρούμε ας πούμε τον εκείνον που έχει αρτοπείο και παραδίδει τα καρβέλια του στη γειτονιά. Βλέπουμε όλο και περισσότερες περισσότερα οχήματα μεταφορικά να αντικαθίστανται. να έχουμε μεγάλα φορτηγά, έχουμε μικρότερα φορτηγάκια και βανάκια που δεν έχουν τον ταχογράφο δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε στο Στρασβούργο. Κάτι που δυσχεραίνει ιδιαίτερα τα πράγματα είναι αυτό. Αν δείτε τι ψηφίσαμε στο πακέτο κινητικότητας, εκεί είδαμε ότι δεν είχαμε πολύ ισχυρή εντολή. Καταφέραμε να περάσει μόλις πριν από τις εκλογές το πακέτο. Αλλά δεν ήταν πολύ ισχυρή εντολή που δόθηκε από το Κοινοβούλιο και αυτό δεν μας βάζει σε ισχυρή θέση όσον αφορά τι διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα στο Στρασβούργο. Για την ομάδα μου είναι όμως σαφές αυτό, Σαφή η κατάσταση και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παλέψει το διάλογο γι' αυτό, στον τριμέρι διάλογο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιονγκέριους, η κυρία Φίντ. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Όταν μιλάμε για ανοιχτό τριμερή διάλογο, ίσως αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν στην τελική τους φάση. Ίσως να μην είμαι πολύ ευγενική έτσι που τα θέτω τα πράγματα, αλλά είναι καλύτερα να τα λέω σαφώς και ξεκάθαρα τώρα και να μην χρειαστεί να τα πω αργότερα. Και να τα λέω αυτά γιατί θα έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες στον τριμερή διάλογο. Ακούω διάφορα μηνύματα εγώ. Ότι αυτή η περίοδος αναφοράς των δύο εβδομάδων δεν στηρίζεται επαρκώς στις διαπραγματεύσεις. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εσφαλμένο. Ξέρω ότι το Συμβούλιο θέλει να επιμηκύνει τις περιόδους αναφοράς, να πάει στις τέσσερις εβδομάδες. Στην πράξη θα καταλήγουμε να έχουμε τρεις ε, μακρές εβδομάδες για τους οδηγούς και μετά μεγάλες περιόδους ανάπαυσης. Ξέρω ότι η συζήτηση ήταν πολύ ζωηρή στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά επιδείνωση των συνθήκων εργασίας των οδηγών, της υγείας τους και τα προβλήματα οδικής ασφάλειας δεν είναι η δική μας στόχη. πρώτερες απόπειρες στο Κοινοβούλιο οι εβδομάδες εργασίας των οδηγών να γίνουν πιο ευέλικτες απέτυχαν. Απέτυχαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από τα τρία χαρτοφυλάκια του πακέτου κινητικότητας, η υποστήριξη του χρόνου ανάπαυσης και οδήγησης ήταν η μεγαλύτερη ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά το τριμερή διάλογο θα έχουμε ξεχωριστές ψηφοφορίες επί των τριών χαρτοφυλακίων και όχι μία ψηφοφορία για το συνδυασμό των χαρτοφυλακίων και ας εν Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει να υπερασπιστούμε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη όταν θα ψηφίζουμε. Ελπίζω λοιπόν ότι είναι σαφές ότι αυτή η περίοδος αναφοράς των δύο εβδομάδων είναι η κόκκινη γραμμή για θετική ψηφοφορία από την πλευρά μας, για θετική ψήφο από την πλευρά μας. Ευχαριστώ. Κυρία Φίντ. Έχετε το λόγο. Μπροστά. Έχετε το λόγο, κυρία Φίντ. Ε, ευχαριστώ πολύ για την όλη παρουσίαση. Θα συνεχίσω στα δανέζικα. 100% θα υποστήριζα τις προειδοποίησεις της κυρίας Ουγγέριος για τις νέες προτάσεις για την παράταση της περίοδου αναφοράς. Κανένα συνδικάτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις τέσσερις εβδομάδες. Αυτή είναι μια σαφής κόκκινη γραμμή. Δεν είναι θέμα μόνο συνθήκων εργασίας για τους οδηγούς των φορτηγών. Αυτή η παράταση, αυτή η επέκταση ε, σχετίζεται και με την οδική ασφάλεια. Την ασφάλεια της κυκλοφορίας για τους οδηγούς, για τους επιβάτες και για τα παιδιά και τους ενήλικες που ίσως είναι στους δρόμους και κυκλοφορούν. Αν το επιχείρημα επέκταση τη περίοδου είναι μεγαλύτερη ευελιξία, η περίοδο αναφορά ε, δύο εβδομάδων δίνει επαρκή ευελιξία, μια αξιοπρεπή ευελιξία. Αν έχουμε την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων για ευελιξία, δίνουμε πολύ μεγάλη ευελιξία για την άθρηση της περίοδου ανάπαυσης σε μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο και ο κίνδυνος είναι στο μέλλον να έχουμε χιλιάδες πολύ βαρέα οχήματα, πολλά βαρέα, βαρέα οχήματα στην Ευρώπη με οδηγούς που θα οδηγούσαν επί τις εβδομάδες χωρίς να έχουν αναπαυτεί και αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάντελ έχει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επενθυμίσω ότι εδώ και μήνες ε, επεξεργαζόμαστε αυτή τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα και ελπίζω να καταφέρουμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Ε, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τον Ντένις ιδιαίτερα για το κείμενο αυτό και εμπιστεύομαι και τα όσα κάνουν και εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω τις βασικές αρχές. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να υπερασπιστούμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια πιο δίκαιη Ευρώπη με συνθήκες εργασίες ε, δίκαιες ε, για όλους τους εργαζομένους ε, στην Ευρώπη, είτε στον τομέα των μεταφορών, είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, αλλά θέλουμε επίσης και ασφάλεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ουσιαστικό σημείο ασφάλεια και εν τέλει συνθήκες εργασίας και άσκησης ενός επαγγέλματος ε, οι οποίοι θα είναι ε, ένομοι και δίκαιοι. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω και δύο-τρία ακόμα ουσιαστικά σημεία επί των οποίων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη φιλοδοξία. Καταρχάς ε, το θέμα των έξυπνων ταχογράφων. Νομίζω ότι επ' αυτού είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν Έξελίξει στην τεχνολογία, αλλά εμείς ως νομοθέτε, θα πρέπει να επιδείξουμε φιλοδοξία και να φροντίσουμε οι ταχογράφοι αυτοί να εγκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, θα ήθελα να πω επίσης ότι όσον αφορά τα ε, ελαφρά οχήματα, θα πρέπει να υπάρξει κάποια πρόοδος, θα πρέπει να μπορέσουμε να καθορίσουμε ένα πλαίσιο, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, διότι αυτή τη στιγμή η οδηγία αυτών των οχημάτων δεν καλύπτονται από καμία νομοθεσία και όσον αφορά τους χρόνους ε, ανάπαυσης ε, και χρόνους ανάπαυσης ε, εντό του θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι πρέπει, θα πρέπει ο χρόνος ξεκούρασης ο εβδομαδιαίος να γίνεται εκτός της καμπίνας του οχήματο, γιατί πραγματικά υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για θέματα ασφαλείας. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ μαζί σας ως προς το γεγονός ότι πρέπει να βρούμε μία λύση για τους οδηγούς που θα είναι εκτός του οδοστρώματος. Εγώ ως σοσιαλίστρια θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε λύσεις για περισσότερη προστασία της ιδιωτικής ζωής των ε, ε, οδηγών και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και ε, βασικό θέμα για τη θητή αυτή. Ευχαριστώ πολύ και για τις ανακοινώσεις ε, στους ε, εισηγητές και περνάμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση και περνάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Και εδώ έχουμε την κυρία Ανδριάννα Σούκοβα. Να σας καλωσορίσω θερμά. A warm welcome and um, you will be... Και δεν ναι, είστε συγγήτρια φυσικά, είστε εδώ για να μας πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα και να σας ε, παρουσιάσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Πρόκειται για παλιά πρόταση, έχει γίνει από το Μάιο πέρσι, αλλά όπως ξέρετε δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων. Επομένως, ε, ε, μπορώ να αφιερώσω χρόνο για να ακούσω τις ιδέες και τις απόψεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε όταν θα καταφέρουμε να διοργανώσουμε τους τριμερείς διαλόγους. Καταρχάς, να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένη που είναι εδώ συγητής, ο κύριος Κάσα, αλλά βλέπω και κάποιους από τους κοιόδης εισηγητές εδώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα κοινό όραμα και ένας κοινό στόχος να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των συνομοθετών των συντομότερων δυνατόν και αυτό είναι μήνυμα το οποίο προέκυψε και από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Οκτωβρίου ότι οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς για τα ταμεία πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο ώστε τα κράτη-μέλη που έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ στις αρχές του 2021 χωρίς καμία καθυστέρηση. Θα ήθελα τώρα να θα αρχαιολογήσω κάποια από τα βασικά στοιχεία τα οποία έχουμε προτείνει. Δεν έχω συνηθίσει να κάνω παρουσιάσει και δεν ξέρω τη διαδικασία. Νόμιζα ότι κάτι λάθος κάνω, ζητώ συγγνώμη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ δυστυχώς δεν φαίνεται καλά η διαφάνεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ περιλαμβάνεται στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο τίτλο του πολιετού μεσονομικού πλαισίου που αφορούν τη συνοχή και τις αξίες. Έχουμε έναν υπότιτλο ο οποίος μπορεί και να φαίνεται εδώ, επενδύουμε στους ανθρώπους και για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ ε, είναι προβεβλημένο όπως θα έπρεπε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και είναι προφανές ότι υπάρχει ουσιαστικό σκέλος του προπολογισμού, το οποίο αφορά ε, κυρίως ανθρώπους. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επίσης είναι τμήμα της ε, πολιτικής συνοχής. Έχουμε κοινό κανονισμό ε, κοινών διατάξεων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και και για την επόμενη προγραμματική περίοδο έχουμε και τα τρία ταμεία τα οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Home ε, το Ταμείο ε, Μετανάστευσης, ε, το Ταμείο για την υγεία επίσης, όλα αυτά καλύπτονται από τις ίδιες διατάξεις. Επίσης, να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημιουργήθηκε το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης και έκτοτε έχει αναλάβει να διευκολύνει την πρόσβαση σε απασχόληση μέσω της κινητικότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσαρμόζονται οι εργαζόμενοι μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ε, συν το χρόνο αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε, αλλά οι βασικοί στόχοι εξακολουθούν να υπάρχουν και εξακολουθούν να ισχύουν. Στην παρούσα περίοδο, μέχρι το τέλος του 2018, μπορώ να σας ενημερώσω ότι έχουμε ήδη υποστηρίξει 26 εκατομμύρια ανθρώπους, από τους οποίους 4,5 εκατομμύρια ήταν από ευάλωτε ομάδες και 3,9 εκατομμύρια ήταν μετανάστες ή ε, από ή αλλοδαποί. Όταν κάνουμε την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, λάβαμε υπόψη τις βασικές ε, γενικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη σήμερα ημέρα, ε, το δημογραφικό, το κλιματικό ζήτημα, τις ε, ιδεολογικές προκλήσεις, ε, δεξιότητες, ε, το επίπεδο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξακολουθεί να είναι απαράδεκτο και οι κοινωνικέ ανισότητε, οι οποίε αποτελούν πλέον ε, σημαντικό σκέλος οποιασδήποτε δράσης, ε, διότι ο κόσμος ε, αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο τη διαφορά μεταξύ των διαφόρων επιπέδων του πληθυσμού και ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο από αυτού του ζητήματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην πρότασή μας έχει στενή σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την πρόταση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Υπάρχουν ε, προκλήσεις πολιτικής, ε, τις οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν όλα τα κράτη-μέλη και προκειμένου να προτείνουμε κάτι το οποίο θα είναι και εύκολο για όλους τους δικαιούχους ε, και θα εξασφαλίσει και συνοχή στην προσέγγιση μας, προτείναμε να συγχωνεύσουμε τα πέντε χρηματοδοτικά μέσα σε ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, λοιπόν, αυτή τη στιγμή καλύπτει για την επόμενη προγραμματική περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την Πρωτοβουλία για την Νεολαία που έχει συγκεκριμένη γραμμή προπολογισμού, το ε, Ταμείο για Ευρωπαϊκή Βοήθεια στους ε, πιο ευάλωτους και στερημένους που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μικρό μεν κονδύλιο αλλά πολύ σημαντικό, Ευρωπαϊκό Μέσο για την Κοινωνική Καινοτομία και το Πρόγραμμα για την Υγεία. Ε, βλέπετε σε σκούρο μπλε έχουμε τα τρία παλιά ταμεία που τώρα είναι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ΣΥΝ ε, και ε, θα υπάρχει συνδιαχείριση. Κυρίως θα γίνεται διαχείριση από τα κράτη-μέλη και τις αρχές των κρατών μελών, ενώ το ε, πρόγραμμα για την κοινωνική καινοτομία και την υγεία θα είναι σε άμεση διαχείριση. το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συν με αυτή τη νέα δομή θέλει να συνδυάσει όλες τις πλευρές πολιτικής ούτω ώστε και τα ταμεία σε κοινή διαχείριση και τα ταμεία σε έμεση διαχείριση να στοχεύουν στους ίδιους στόχους. Όλοι λοιπόν θα συμβάλλουν σε αυτή την ε, επίτευξη των κοινών στόχων. Θέλουμε να υπάρχει συνέχεια. Οπότε το τμήμα απασχόλησης και κοινωνικής καινοτομίας του Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ θα καλύπτει τα υπάρχοντα προγράμματα, τους δύο άξονες των υπαρχόντων προγραμμάτων και τα άλλα που είναι η μικροχρηματοδότηση και άλλα θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και στο InvestEU. Θα έχουμε εκεί επενδύσεις για τις κοινωνικές δεξιότητες. Και εκεί θα πάει και η διευκόλυνση, την κινητικότητα. Για να υπάρχει συνέχεια, επειδή έχουμε πολλές δοκιμές και πειραματισμό στους διάφορους τομείς κοινωνικής πολιτικής, θα αξιοποιήσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτών των πειραματισμών να αποτελέσουν τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα για τη δράση των κρατών μελών. Ο προπολογισμό που προτείνουμε είναι 101,2 δις εκ των οποίων 100 δισεκατομμύρια θα είναι υπό ε, κοινή διαχείριση και οι ακραίως ε, περιφερειακές περιοχές, απομακρυσμένες περιοχές και οι περιοχές με χαμηλό πληθυσμό θα πάρουν 400 εκατομμύρια. Και για να ενθαρρύνουμε την διεθνή συνεργασία δώσαμε 200 εκατομμύρια. Για ένα συγκεκριμένο στόχο εντό εντός της πλευράς κοινή διαχείρισης. Και το τμήμα υπό άμεση ή έμεση διαχείριση θα περιλαμβάνει απασχόληση και κοινωνική καινοτομία 761, ενώ η υγεία είναι μόνο 413 εκατομμύρια. Στοχεύουμε επίσης να υπάρχει ευελιξία και δυνατότητα τα κράτη-μέλη να προωθούν προγράμματα με βάση τους συγκεκριμένους στόχους του Ταμείου για να αντιμετωπίσουν τις ειδικέ προκλήσεις σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Επίσης θα υπάρχει στενότερη σχέση μεταξύ του Ταμείου αυτού και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και αυτό φαίνεται και στην προετοιμασία των ε, καταχώρα εκθέσεων για το 2019. Υπάρχει ένα παράδειγμα που ε, αφιερώνεται ειδικά σε αυτό. Εκεί εκφράζει η Επιτροπή έναντι κάθε κράτους μέλους την άποψή της για το ποιες είναι οι κύριες ε, προκλήσεις και τα κενά επενδύσεων που έχουμε εντοπίσει και προτάσεις της Επιτροπής πού ε, μπορούν να πάνε οι ευρωπαϊκοί πόροι για να κλείσουν αυτά τα κενά. Το παράρτημα αυτό είναι η βάση για το διάλογο με τις ε, διαχειριστικές αρχές που ετοιμάζουν τα έγγραφα προγραμματισμού τους για την επόμενη περίοδο. Στο κανονισμό για το esf sin υπάρχει σαφής απέτηση η συστάση αναχώρα που βγαίνουν από τις εκθέσεις αναχώρα να αναφέρουν τις προτεραιότητες των, στα πλαίσια του ESFC ούτως ώστε να δούμε πώς θα γίνεται η κατανομή των πόρων για να βοηθήσουμε έτσι καλύτερα τα κράτη-μέλη να κάνουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Και επίσης έχει και περιφερειακή διάσταση η αξιολόγησή μας και η ανάλυση πολιτικών, ώστε τα κράτη-μέλη που έχουν ε, διαχείριση αναπεριφέρειας να έχουν ε, σαφή διαφοροποίηση, διαφοροποίηση με βάση τις ανάγκες των διαφόρων περιοχών. Έχουμε πολύ λίγες απαιτήσει για συγκέντρωση ανά ε, θεματικό τομέα, τρεις συγκεκριμένοι. Πρώτα απ' όλα. Ένα πολύ θαραλέο βήμα. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη να αφιερώσουν τουλάχιστον 25% για μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Εδώ είχαμε 20% ως απέτηση, για το, στην προηγούμενη περίοδο δηλαδή, για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και κατά την τρέχουσα περίοδο ήδη αφιερώσαμε 24%. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν αυτές οι κοινωνικές προκλήσεις στα κράτη-μέλη και υπάρχει σημαντικός σημαντική σύνδεση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικού Δικαιωμάτων και της ανάγκης ακριβώς να αποδίδονται τουλάχιστον 25% για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού. Πρέπει να μειωθεί ε, το επίπεδο της φτώχειας, να στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες, ούτω ώστε ε, οι μειονεκτούσες ομάδες και οι μειονότητες να συμπεριλαμβάνονται στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας. Πρέπει να γίνουν περισσότερα εδώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βοήθεια για τους ε, πιο μειονεκτούντες πρέπει οπωσδήποτε να λάβει το 2%. Τουλάχιστον το 2% από τους πόρους του esf sin Υπάρχει ακόμη ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το Ταμείο αυτό. Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένη απτή στήριξη στα άτομα αυτά, αλλά και συνοδευτικά μέτρα συμβουλές, ε, κοινωνικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία ή να επανενταχθούν. Και η ενδιάμεση αξιολόγησή μας έδειξε ότι τα καταφέρνουμε. Αυτό το ταμείο λοιπόν για τους πιο μειονεκτούντες έχει βοηθήσει πολλά άτομα στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να πω ότι τουλάχιστον 30% από τους ε, ωφεληθέντες είναι παιδιά. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η στήριξη. Θέλουμε να τους αποδώσουμε 3,8 δις κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Αυτό το minimum 2% σημαίνει 2 δις. Αλλά ήδη στις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη ξέρουμε ότι ορισμένα θέλουν να πάει το 7-8% από τη χρηματοδότηση του ESFC. Προ τα άτομα αυτά τα πιο μειονεκτούντα με διαφορετικούς τρόπους να τα στηρίξουν. Τώρα, η απασχόληση των νέων. Επίσης μας απασχολεί. Κάνουμε πρόταση γι' αυτό. Η ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επίγον θέμα σε πολλά κράτη-μέλη. Εμείς προτείναμε ότι οι νέοι need που είναι δηλαδή ούτε σε εκπαίδευση, ούτε κατάρτιση, ούτε απασχόληση, δηλαδή μεταξύ 15 και 29 ετών, είναι 12-9% στα κράτη-μέλη. Άρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα με βάση την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Προτείνουμε τα κράτη-μέλη, όπου τα επίπεδα των ατόμων αυτών NEET είναι υψηλότερα από τον ε, μέσο όρο, τα κράτη-μέλη λοιπόν αυτά θα πρέπει να αφιερώσουν τουλάχιστον 10% από το, τους πόρους του ESF-SYN για τα άτομα αυτά, για τους νέους αυτούς. Οι τελευταίες μας εκθέσεις τέλη του 2018 αποδεικνύουν ότι το πρόγραμμα αυτό βοήθησε 3,5 εκατομμύρια νέων στην Ευρώπη. Είναι υποχρέωση των κρατών μελών. Ενώ η πρωτοβουλία για τους νέους στήριξε μόνο 20 κράτη-μέλη όπου είχε, είχαμε πολύ ψηλά επίπεδα ανεργίας νέων. Με αυτή τη χρηματοδότηση μέχρι τέλος του 2018 έχουμε ήδη στηρίξει 2,7 εκατομμύρια νέους. Τους βοηθήσαμε να βρουν εργασία ή να κάνουν κάποια μαθητεία, κάποια κατάρτιση ή συμπληρωματική εκπαίδευση και δεξιότητες. Την επόμενη περίοδο, χρησιμοποιώντα τα τωρινά στατιστικά στοιχεία, θα έχουμε νέα κράτη-μέλη, τα οποία θα είναι υποχρεωμένα να διατηρήσουν το ελάχιστο 10% της απασχόλησης Βουλγαρία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρος, Ρουμανία, Σλοβακία και Κροατία. Θα ενισχύσουμε την πολιτική και το πλαίσιο για την ε, απασχόληση των νέων. Αυτή ήταν μια δέσμευση που ανέλαβε η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από μερικούς θα συζητήσουμε και μαζί με εσά και με διάφορους εκπροσώπους ε, οργανώσεις των νέων πώς να κάνουμε τις τέσσερις προσαρμογές και πώς να εξασφαλίσουμε ότι τα μέτρα αναπτύσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι οι νέοι γρήγορα, γρήγορα να την χάνουν τη σωστή ε, υποστήριξη. Τώρα, στα πλαίσια του 25% για την συμπερίληψη και την υποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συμπεριλάβουμε και τη φτώχεια των παιδιών. Συμφωνούμε το Κοινοβούλιο ότι αυτά είναι θεμελιώδη μέτρα που απαιτούνται για τη μελλοντική ευημερία των παιδιών και για θετική ανάπτυξη των παιδιών. Η ευημερία των παιδιών είναι η αρχή υπαριθμών 11 του κοινωνικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και συμπεριλαμβάνεται στις στάσεις αναχώρα για κάποια κράτη-μέλη στις σχετικές εκθέσεις αναχώρα. Βασίζουμε τις προτάσεις μας στις εκθέσεις αναχώρα και τις σχετικές συστάσεις επί των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επενδύσεις για τα παιδιά και διάφορα μέτρα ήδη έχουν εφαρμοστεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο για να καλύψουμε τα παιδιά, να τους δώσουμε πρόσβαση σε ε, μέρημνα και σε παιδεία, μέτρα για κοινωνική συμπερίληψη των οικογενειών τους, και αρκετά σημαντικά ποσά θα τεθούν αν εφαρμοστούν σωστά οι αναχώρα συστάσεις και αυτή η σωστή εφαρμογή του προγράμματος θα υποστηρίξει θέματα παιδείας σε 10 κράτη-μέλη, πρόσβαση στην παιδική μερίμνα σε 5 κράτη-μέλη και πρόσβαση στην υγεία σε άλλα 5 κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να το υπογραμμίσω αυτό, διότι υπάρχει αύξηση ζήτησης όσον αφορά δυνατότητες χρηματοδότησης τομείς που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και έχουμε περιορισμένο κονδύλι για το ταμείο αυτό και συγκεκριμένους στόχους που έχουν προταθεί και θα πρέπει να είμαστε πολύ εστιασμένοι όσον αφορά τις δαπάνες και τους στόχους. Θέλουμε θεματική προσέγγιση να αντιμετωπίσουμε τις δυσχερέστερες καταστάσεις στα κράτη-μέλη. Όχι μια γενική προσέγγιση, θέλουμε να πετύχουμε σημαντική αλλαγή στις καταστάσεις και όχι εμβαλωματικές λύσεις. Υπάρχει μια οριζόντια αρχή που μας ενδιαφέρει. Είναι η σύμπραξη, η συνεργασία. Θέλουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε σχετικέ διατάξεις για τι εργασίες στο σχετικό κανονισμό με τι εφαρμοστικές διατάξεις. Οπότε είναι προπόθεση για τη χορήγηση πόρων από όλα τα ταμεία για το ESF συν. Έχουμε συγκεκριμένη διάταξη και ζητούμε από του εμπλεκομένου φορείς να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δυναμικό όταν εμπλέκονται στην υλοποίηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ESF συν. Θα σταματήσω εδώ. Θέλω να ακούσω τις δικές σας απόψεις, προτάσεις, πριν ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να σας τα παρουσιάσω αυτά. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, κυρία Αντριάννα Σούκοβα. Πριν ξεκινήσουμε με τους ομιλητές, να σας πω ότι η κυρία Σιμώνα Μπαϊντασάρ έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Είναι εδώ? Όχι, ναι. Α, δεν είναι εδώ. Αν τα γενέθλιά της σήμερα. Καλώς, συνεχίζουμε. Ντάβιτ Κάσα, ο εισηγητής και μετά θα μιλήσουν οι σκιώδεις. Ο κύριος Ράνκε, να ξεκινήσει, η κυρία Ράνκε. Ας ξεκινήσει πρώτη, γιατί πρέπει να φύγει. Μετά τον κύριο Κάζα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Σούκοβα για την παρουσίαση που έκανε. Σωστά αναφέρθηκε στη σημασία του κοινωνικού ταμείου. Είναι να συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη της Ρώμης. Από την αρχή έγινε αντιληπτή η σημασία του ταμείου. Είχε σημασία για την Ενωμένη Ευρώπη. Και οι ανάγκες του 57 είναι διαφορετικές από τις σημερινές. Σήμερα έχουμε διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές προκλήσεις, άρα χρειαζόμαστε σύγχρονες ιδέες για να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε ότι στο άθρο 70 αναφερθήκαμε διατίθεται πόροι για την επίτευξη των στόχων για την εγγύηση των για τα παιδιά. Είναι κρίσιμο αυτό για τα παιδιά και για την εκλεγήσα πρόεδρο που ανέλαβε κάποιες δεσμεύσεις να προωθήσει το μέσο αυτό εγγύησης για τα παιδιά. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την προσέγγιση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και αν υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σχετίζονται με τους στόχους της εγγύησης για τα παιδιά θα ήμασταν πολύ ευτυχείς αν μπορούσατε να μας πείτε αυτές τις απόψεις σας. Μετά, το δεύτερο ερώτημα αφορά και ένα πρόβλημα. Σχετικά με το άθρο 7, το Κοινοβούλιο ανησυχεί για τη συμπερίληψη του άθρου 7 που τη συμπεριέλαβε το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις είναι, δίνει, προβλέπει περιορισμένο χρόνο για τη συζήτηση σημαντικών θεμάτων. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με αυτή την ατυχή συμπερίληψη των λόγω άρθρου. Ευχαριστώ κύριε Κάζα. Η Σκιώδης τώρα. Η κυρία Ράιντκε, ο κύριος Μονιφέη, η κυρία Σεμέδο, η κυρία Μπαλτασάρ, Κύριε Ραφαέλτσκα και κύριε κυρία είναι στον κατάλογό μου για τους και ηγητές. Κύριε Ράντκε, έχετε το λόγο. Κυρία Ράντκε. Θα είμαι πολύ γρήγορη. Ευχαριστώ που αλλάξατε κάπου, κάπως τους όρους στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να φύγω. Τρία σημεία να θίξω που πιστεύω ότι θα είναι και τα καυτά θέματα. Ο κ. Κάζα αναφέρθηκε σε κάποια αυτά το θέμα του όγκου πήραμε μια θέση ότι θα χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και θα επιμείνουμε από αυτού και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια τη συναπόφαση, να συζητηθεί στου τριμερεί διαλόγου και πρέπει να είμαστε πολύ στεναροί στη θέση μα. Το ίδιο ισχύει και για την προσημείωση του earmarking. Είπατε ότι ήδη έχετε φιλόδοξη πρόταση με το 25%. Εμείς το ξεπερνάμε ακόμα αυτό και το κάνουμε αυτό για λόγους που έχουμε. Αν δούμε την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για θέσεις εργασίας, να μιλήσουμε για απασχόληση, αλλά κοινωνική ένταξη, κοινωνικά θέματα, κυρίως σε εκπιοχές που ενισότητες στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται, αυτά τα χρήματα χρειάζονται πάρα πολύ και το ίδιο ε, χρειάζεται, είπατε 2%, ελάχιστες δαπάνες, έχουμε 3% και θα επιμείνουμε από αυτούς στους τριμερείς διαλόγους. Είναι σημαντικό επίσης οι πιο στερημένες ομάδες στην κοινωνία μας να μπορούν να ωφεληθούν από αυτά τα χρήματα. Τέλος, να αναφέρω κάτι το οποίο νομίζω ότι όταν μιλάμε στους δικαιούχους και με τον κόσμο που τα έρχονται σε επαφή με τα χρήματα πάντα μας το λένε ότι πρέπει να λαχιστοποιήσουμε το διοικητικό άχθος για τους διάφορους οργανισμού, διότι θέλουμε να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για την κοινωνία των πολιτών όχι μόνο για του μεγάλους φορεί, που έχουν διοικητικό προσωπικό. Στου τριμερεί διαλόγου θα πρέπει να εστιαστούμε από αυτού και καλό και όλου του συναδέλφου εδώ να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιβαρύνουμε πολύ του οργανισμού στην υλοποίηση των μέτρων. Και τέλο, μια έκκληση απευθύνω σε εσά και σε όλου μα και κυρίω σε όσου πηγαίνουμε στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Νομίζω ότι ήδη πραγματικά δεν μα μένει πολύ χρόνο. Θα πρέπει να έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Διότι αν δούμε τι διαφορέ θέσει που υπάρχουν, υπάρχουν διαφωνίε. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε το θέμα δεν θέλω να έχουμε ένα μεγάλο κενό όσον αφορά τη χρηματοδότηση των διαφόρων φορέων, διότι η δουλειά που κάνουν είναι πάρα πολύ αναγκαία. Με αυτή την έκκληση θα σταματήσω και λυπούμε πρέπει να αποχωρήσω και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σε μεταγενέστερο στάδιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη δήλωσή σας. Ο κύριος Μπράντο Μπενιφέη έχει το λόγο τώρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσία της εδώ, κυρίως ε, την κυρία Ανδρέα Νασούκοβα λοιπόν για την παρουσίαση και τους συναδέλφους ε, και για κάποιους νέους συναδέλφους που προφανώς δεν μπορούσαν να παρακολουθούν βήμα-βήμα τα όσα έχουν γίνει από την προηγούμενη θητεία. Νομίζω ότι έτσι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων εν ώψη και του τριμερούς ε, διαλόγου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, το οποίο εντός ολίγου θα ξεκινήσουμε με μια ευαίσθητη διαπραγμάτευση. Επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Νταβίτ Κάσα ε, τον συγητα μας, ο οποίος ε, έχει το δύσκολο έργο να υπερασπιστεί τη θέση που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που όπως υπενθυμίσαμε ήδη είναι μια πάρα πολύ ε, φιλόδοξη θέση και ο βασικός στόχος είναι να αναγνωριστεί το βασικό μέσο για την συγκεκριμένη εφαρμογή ενός σημαντικού σκέλους ε, του κοινωνικού θεματολογίου και την υλοποίηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των ε, Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Υπάρχουν ε, απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και προσεγγίζει την Ευρώπη στους πολίτες. Ελπίζουμε λοιπόν να εργαστούμε καλά όλοι, όλη η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και ο συζητητής για τους Σοσιαλιστέ και δημοκράτε Είμαι περήφανο ε, που συνέβαλα στην ενίσχυση του κειμένου, παρουσιάζοντας μια σειρά από τροπολογίε κυρίως στο θέμα της εργασίας και της κατάρτισης, της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πέρα από την γενικότερη αναδιοργάνωση του κοιμώνου και των συγκεκριμένων στόχων, ε, τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Κοινοβούλιο προτείνουμε επίσης να εντείνουμε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ε, ανεργίας των νέων. Ο στόχος είναι να μετατραπεί η λεγόμενη πρωτοβουλία για την ε, απασχόληση της νεολαίας, τη λεγόμενη Youth Initiative, για να αντιμετωπίσουμε και κάποιες ε, απρόβλεπτες κρίσεις ε, στον τομέα της απασχόλησης, όπως αυτά τα οποία διαπιστώσαμε στα χρόνια της κρίσης. Επίσης, θεωρήσαμε απαραίτητο να αυξήσουμε τα διάφορα ποσοστά της θεματική συγκέντρωση του άρθρου 7, για να δοθούν σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης, ε, στο Ταμείο για τη Βοήθεια προς τους ε, ε, της πιο μειονεκτικής ομάδας. Ε, θέλουμε να υπερασπιστούμε και το πρόγραμμα ΦΕΑΤ και να συμπεριληφθεί στο νέο ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, αλλά να λαμβάνει και κατάλληλη χρηματοδότηση και υποστήριξη, ώστε οι πάρα πολλέ οργανώσει που παρέχουν βοήθεια σε αυτού που την έχουν περισσότερη ανάγκη να μπορούν να δραστηριοποιούνται καταλήλω. Χαίρομαι που ο πρόεδρο Σασόλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστήριξε δημόσια αυτό το θέμα ε, και υποστήριξε και το έργο που έκανε το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε σημείο συνάντηση με το Συμβούλιο σε αυτό το λεπτό σημείο. Θέλαμε επίσης ε, να υποστηρίξουμε και άτομα με αναπηρία, διότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την εργασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θέλουμε το νέο κοινωνικό ταμείο να συγχρηματοδοτήσει και ε, εθνικά σχέδια για τη μετώπιση της ε, φτώχειας και επιδόματα για το ε, εισοδήματα και επίσης ε, θέλουμε να έχουμε μια πιο άμεση πρόσβαση για τοπικές αρχές και οργανώσεις του, του τρίτου τομέα για να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα ένταξης σε τοπικό επίπεδο. Ε, το Κοινοβούλιο είχε ήδη εκφράσει την άποψή του στην έκθεση πρωτοβουλία για την ένταξη των μεταναστών. Εγώ ήμουν εισηγητή επί του θέματο πριν από κάποια χρόνια και θελήσαμε να προτείνουμε και ένα νέο πρόγραμμα, την εγγύηση για τα παιδιά, που θα επιτρέψει σε πολλά παιδιά που προέρχονται από μειονεκτικέ οικονομικέ και κοινωνικέ συνθήκε να έχουν πρόσβαση σε ουσιαστικέ υπηρεσίε. Χαίρομαι που η πρόεδρο Φόντερ Λάιεν ε, οικειοποιήθηκε την πρόταση ω ε, υποψήφια πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν επιβεβαιωθεί θα διαδραματίσει ένα πάρα πολύ δραστήριο και θετικό ρόλο κατά τη διαπραγμάτευση και για αυτό το σημείο. Και νομίζω ότι από αυτού θεωρούμε ότι έχει αλλάξει και ο προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίσως. Ε, φαίνεται να υπάρχει ε, διαφορετική στάση γιατί ήταν μεγαλύτερη η δισταγμή τους ε, στο παρελθόν. Και έλος θα ήθελα να κάνω κάποιες επικρίσεις. Καταρχάς δεν κρύβω ότι ανησυχώ ε, για το βασικό στοιχείο. Υπάρχει ένα πολύ σύνθετο θέμα το οποίο έχει μεγάλη σχέση και με άλλα θέματα διαπραγμάτευσης, κυρίως το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις, το CPR. Ελπίζω να μπορέσει να ξεκινήσει το συντομότερα δυνατόν ο τριμερής διάλογος ως να μην καθυστερήσει η συζήτηση για ένα τόσο λεπτό ζήτημα. Θέλουμε η επόμενη προγραμματική περίοδο να ξεκινήσει εγκαίρω και πολύ σημαντικοί πόροι όπω οι πόροι του Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ ε, δεν πρέπει να καθυστερήσουν γιατί θα καθυστερήσουν οι διαπραγματεύσει. Είμαστε βέβαιοι ότι εμεί ω Κοινοβούλιο θα κάνουμε αυτό που τη αναλογεί και νομίζω όμω ότι δεν θα είμαστε διατεθειμένοι και ήταν σαφώ και ο εισηγητή ω προ αυτό. Δεν θα θυσιάσουμε την ποιότητα των θεμάτων ε, λόγω ε, χρόνων οι οποίοι μπορεί να είναι απαγορευτικοί ή να θεωρηθούν κάποια θέματα επίγοντα. Απλώς και μόνο για να επιτευχθούν κάποιοι πολιτικοί στόχοι. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε σύντομα τους τριμερείς διαλόγους για να αποφύγουμε τέτοιες ε, περιπτώσεις. Και μια δεύτερη επίκριση, το ακούσαμε ήδη, θέλω να το επαναλάβω κι εγώ, το λεγόμενο αένο θέμα των negotiating boxes. Ε, το Κοινοβούλιο θα θελήσει να συζητήσει και τα θέματα του κανονισμού και τι διάφορε θεματικέ ενότητε. και υπάρχουν συγκεκριμένε αλλαγέ στη δομή του προγράμματο και σε επίπεδο προγραμματισμού και υπάρχουν και κάποιε πτυχέ οι οποίε είναι αμυγό χρηματοδοτικέ. Πρόκειται για βασικά στοιχεία τα οποία αφορούν τη συνήθι νομοθετική διαδικασία και τη συναπόφαση που πρέπει να συζητηθούν στον τριμερό διάλογο και ελπίζουμε να υπάρξει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σημεία αυτά. Ευχαριστώ για την προσοχή σα και καλή δουλειά σε όλους werde auf Deutsch Herzlichen Θα συνεχίσω στα γερμανικά. Ευχαριστώ. Τον προηγούμενο ομιλική, ομιλητή. Και τώρα η κυρία Μόνικα Σεμέδο από το Renew, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ γερμανικά μιλάω. Ευχαριστώ την κυρία Σούκοβα για την παρουσίαση του ESF-SYN. Η καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Τα έχει πάει καλά. Έχει σημειωθεί πρόοδος. Αλλά πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στην απασχόληση των νέων. 10% των πόρων πρέπει να πάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την πρωτοβουλία για τους νέους. Εμείς του ΡΙΝΙΟΥ και το Κοινοβούλιο απαιτεί 15%. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε για να το επιτύχουμε. Όσον αφορά την εγγύηση για τους νέους και για την ε, διαβίου κατάρτιση πρέπει να γίνουν περισσότερα και να συμπεριληφθούν και οι μετανάστες. Η μετανάστευση είναι μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να βοηθήσουμε του συμπολίτε μας αυτούς που είναι τμήμα της κοινωνίας μας και θα είναι τμήμα και της μελλοντική μας κοινωνίας να του βοηθήσουμε να ενταχθούν. Τώρα να έρθουμε στα άτομα που έχουν, ε, μάλλον συγγνώμη, στο EFRD, το Περιφερειακό Ταμείο, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που χρειάζεται τα περισσότερα. Πρέπει οπωσδήποτε ε, να υπάρξουν μέτρα εδώ και για τους μετανάστες να αξιοποιήσουμε τα, τους πόρους αυτούς μακροπρόθεσμα. Και μια συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά την απλούστευση και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Πώς ε, θα γίνουν αυτά συγκεκριμένα στην πράξη. Διότι πολλές φορές περιμένει κανείς μήνες για να λάβει τα χρήματά του διότι δεν υπάρχουν πόροι και πρέπει να πάρουν αποθεματικά. Πώς είναι δυνατόν αυτό. Θα πρέπει όταν ξεκινάει ένα πρόγραμμα να γίνονται σύντομα οι πληρωμές. Βεβαίως, ε, ε, μέσω της ευελιξίας θα πρέπει να αποφύγουμε και την ε, καταχρηστική χρήση αυτών των πόρων. Ευχαριστώ κυρία Σεμέντο. Η κυρία Μπαλντασάρε. Α, δεν είναι παρούσα. Δεν είναι εδώ. Η κυρία Ραφάλσκα, ECR. Ευχαριστώ, θα μιλήσω πολωνέζικα. Και θα ήθελα καταρχάς να ευχηθώ χρόνια πολλά στη συνάδελφο που έχει τα γενέθλιά της. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, τις πολύ ενδιαφέρουσες που μας δόθηκαν. Αυτές καταδεικνύουν τη δυσκολία των διαπραγματεύσεων που μας περιμένουν. Είναι τεράστιο το θέμα που συζητούμε. Μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Αυτή η πτυχή ΣΥΝ ε, έχει επιρροή όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα στην Πολωνία. Ξέρουμε διάφορα προγράμματα που έχουν αυτό το συν. Εκεί προβλέπονται συμπροματικοί πόροι για τα κοινωνικά θέματα. Και σε επίπεδο ευρωπαϊκό βλέπουμε ότι έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ που διευρύνει κατά κάποιο τρόπο το πεδίο δράσης. Υπάρχει ζήτηση όσον αφορά τις πλέον ευάλωτε ομάδες. Κάποιοι είπαν να δοθεί 3% και όχι 2% για τις πλέον ευάλωτε ομάδες, αλλά πρέπει να προσέξουμε μια άλλη πτυχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή αφορά την αποτελεσματικότητα των δαπανών, των πόρων που διατίθενται. Πρέπει να υπάρχουν πόροι για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων, παραδείγματος χάρη αλλά τα προγράμματα τα σχετικά για την απασχόληση των νέων έχουν δρομολογηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δαπανούνται χρωστά, σωστά τα χρήματα. Μετά μιλάμε για την εγγύηση για τα παιδιά. Αν θέλουμε αυτή η εγγύηση για τα παιδιά πραγματικά να έχει αποτελέσματα, χρειαζόμαστε σωστά ισχυρά μέτρα δεν μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό το τομέα και να εφαρμόσουμε πολιτική με μικρά βήματα. Αλλιώς θα μας επικρίνουν και θα μας πούν ότι δεν εφαρμόζουμε σωστές πολιτικές για να βοηθήσουμε τα παιδιά, τους νέους ή ε, τις πολυμελείς οικογένειες. Και κάτι άλλο. Στο κείμενο γίνεται λόγος ε, για κοινωνική οικονομία που συμπεριλαμβάνεται σε συγκεκριμένο στόχο και έχω μία ερώτηση η οποία αφορά το θέμα αυτό. Η συμπερίληψη των κοινωνικών επιχειρήσεων σε έναν ειδικό στόχο δεν θα περιθωριοποιήσει ε, κάποιους ε, στα πλαίσια της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, τους φορείς εκείνους που ασχολούνται με την κοινωνική οικονομία. δεν έχουν πάντα μεγάλη εμπειρία. Σε κάποιες χώρες δεν έχουν και μακρά εμπειρία, όπως σε άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Όσον αφορά την Πολωνία, έχουμε φορείς στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της αλληλεγγύης, αλλά αυτοί, οι φορείς, αυτοί οι οργανισμοί μας λένε ότι να συμπεριληφθούν αυτά, αυτή οι στόχη σε ειδικό στόχο μπορεί να αποδυναμώσει τις σχετικές δράσεις που εφαρμόζονται. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ραφάλσκα. Τώρα κανονικά θα έπρεπε να μιλήσει ο κύριος Γκουσμάου. Αλλά δεν τον βλέπω. Οπότε να περάσουμε στις ομιλίες ε, των άλλων συναδέλφων. Πάτον, Ντόμπρεφ, Ζάντερ, Μάντερ και Σατούι. και μετά και ίσως και άλλοι. Ο κύριος Πάτσαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Είναι ένα τομέα που με ενδιαφέρει πολύ. Πριν είχα τη, να έχω την τύχη να είμαι βουλευτή, ασχολούμουν με φιλανθρωπικού οργανισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω μεγάλε επιφυλάξει και θέλω να με διαφωτίσετε. Η παρουσίασή σα εστιάστηκε επί διαδικασιών και γραφειοκρατίας και όχι τόσο επί επιδόσεων του Ταμείου. Και αν δούμε το όλο ιστορικό του Ταμείου, οι επιδόσει ήταν αρκετά απογοητευτικέ μέχρι τώρα. Ένα στου τέσσερι Ευρωπαίου ζει στη φτώχεια σήμερα. Η ανεργία των νέων, όπω στην Ελλάδα, είναι στο 40%. Άρα ανησυχώ πολύ. Πριν προχωρήσουμε και δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα για το πρόγραμμα, να δούμε πώ καλύτερα μπορεί να αποδώσει επένδυση. Σωστά αναφερθήκατε στη θεματική συγκέντρωση και όχι εμβαλωματική προσέγγιση. Κάπως έτσι το παρουσιάσατε. Βλέποντας τα έγγραφα που υπάρχουν και το κείμενο αναφέρονται τρία θέματα, 11 στόχοι και ε, πάρα πολλοί τομεί στους οποίους θα αναπαθούν τα χρήματα. Πρέπει να δείτε δύο πράγματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, χρειάζεται σοβαρή δέσμευση παρακολούθησης και αξιολόγηση, πραγματικά σοβαρή, χρειάζεται να παρακολουθούμε όλη την αλυσίδα. Πριν καν ξεκινήσει το πρόγραμμα να ξεκινά ο έλεγχος, για να μπορούμε να κρίνουμε καθημερινά, κάθε, και κάθε χρόνο, κάθε τρία χρόνια, κάθε πέντε χρόνια την ε, επιτυχία. Αποτελέσματα. Αναφερθήκατε στα 2,7 εκατομμύρια νέους που βοήθησε το Ταμείο να βρουν απασχόληση. Η ερώτησή μου, οι νέοι αυτοί έχουν ακόμα δουλειά, είναι ακόμα στην παιδεία, βγήκαν από τη φτώχεια, τους βοήθησε. Αυτές τις πληροφορίες χρειαζόμαστε. Το δεύτερο. Λέγαμε ότι θα απλουστευτούν οι διαδικασίες μέσω του ESF ε, ε, συν ε, και τα πέντε ταμεία έγιναν ένα και αυτό δείχνει μια πλούστευση θεωρητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο. Επιτόπου τι γίνεται. Προσωπικά ξέρω ότι για, τα, για μικρότερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς που είναι στην πρώτη γραμμή και κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά μακροπρόθεσμα είναι οι φορείς εκείνοι που ε, δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση από αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ δύσκολο να έχουν πρόσβαση. Τι θα κάνετε για να διευκολύνετε αυτούς τους μικρότερους οργανισμούς. Πριν σπαταλήσουμε περισσότερα χρήματα, εγώ θα έλεγα ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση και η μείωση της γραφειοκρατίας είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πάτεν. Η κυρία Ντόμπρεφ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, είμαστε μια από τι πιο αναπτυγμένε περιοχέ του κόσμου και μία από τις ισχυρότερες οικονομίες και έκανε πολλά η Ευρώπη μέσω της ενιαίας αγοράς, με τις πολιτικές συνοχής, ε, με την ΟΝΕ και τα λοιπά για να φτάσει σε αυτό το σημείο ένωση. Επειδή ζούμε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο οικονομικά ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου, είναι πολύ λυπηρό να διαπιστώνουμε ότι έχει αυξηθεί ανισότητα την τελευταία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Ναι μεν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο που αντελήφθησαν κατά την ε, προηγούμενη θητεία την ε, επίγουσα κατάσταση αυτή και χαίρομαι που βλέπω και ότι και από το ΕΛΚ και οι σοσιαλδημοκράτες, οι πράσινοι, το ΡΙΝΙΟΥ όλοι αυτοί βλέπω ότι συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις για να χρηματοδοτηθεί περισσότερο η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η ισχυρή Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή και μείωση των ανισοτήτων. Και ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά βεβαίω χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοδότηση τη κοινωνική πολιτική. Δι χρημάτων. Αλλά η και αποτελεσματικότητα είναι σημαντική. Και αμφισβητήθηκε τα τελευταία χρόνια. Γιατί τα πολλά χρήματα, αλλά σε κάποια κράτη-μέλη η ανισότητα έχει αυξηθεί, καθώς και η ανισότητα μεταξύ κρατών μελών. Οπότε, θα αρκέσουν οι πόροι. Θα έχουν δυνατότητα να παρακολουθούμε, αλλά και να παρεμβαίνουμε να διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε κάποια κράτη-μέλη δεν είναι αποτελεσματικές. Ξέρω ότι έχουμε τις αιτήσει αξιολογής κτλ. Αλλά θεωρώ ότι δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς που να μας επιτρέπουν να παρεμβαίνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται δεν αρκούν ή δεν κάνουν αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουν ή απλώς δαπανούν πολλά χρήματα για πενιχρά αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν όλοι μαζί, Επιτροπή Κοινοβούλιο και ελπίζουμε και το Συμβούλιο, να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορούμε να ελέγχουμε και να παρεμβαίνουμε πολύ ταχύτερα και πολύ πιο αποτελεσματικά κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντόμπρεφ, λοιπόν, να διορθώσουμε τώρα το κατάλογο. Θα κάνουμε μία αλλαγή. Τώρα η κυρία Πισλάρο, Ζάντερ, μετά Λάντερ, μετά Σατούρι. Και νομίζω ότι έτσι θα καταλήξουμε. Ο κύριος Πισλάρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Επίσης πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις από πλευράς μου και πολύ σύντομα σχόλια. Καταρχάς αναφέρεστε στη σημασία που προσδίδουμε τη σήμερα ημέρα στα παιδιά και τα στερημένα παιδιά κυρίως. Εξετάζουμε την πρόταση για τις πρώτες 100 ημέρες της Προέδρου Ούρσουνα Φόντερ Λάιεν για την εγγύηση για τα παιδιά. Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για το πώς σκοπεύετε να ε, εντάξετε το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και να δώσετε χώρο στο θέμα αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η εγγύηση για τα παιδιά δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο για την εφαρμογή. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε τη στέγη, τη διατροφή και την εκπαίδευση και όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν σε επίπεδο κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ότι ο ολοκληρωμένος τρόπος είναι κάτι προς εξέταση ως τρόπος εφαρμογής ε, στις ε, συστάσεις αναχώρα και ούτω καθεξής, αλλά έχετε προσεγγίσει καθόλου το θέμα. Σε τι αποτελέσματα έχετε καταλήξει από την αξιολόγηση που γίνεται για την ε, ε, εγγύηση για τα παιδιά και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Ε, τώρα, το θέμα της ασφάλειας. Δεν αναφέρομαι τόσο περισσότερο στο θέμα της απλοποίησης, αλλά την εξέλιξη των κοινωνικών υπηρεσιών παγκοσμίω. Τη σήμερα ημέρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο προχωρά από το πρώτο βήμα της, την εσωτερήκευση των υπηρεσιών στο επόμενο βήμα εξωτερήκευση των υπηρεσιών και πάμε και προς ένα σύστημα το οποίο δίνει συμβάσεις για κοινωνικά αποτελέσματα και ένα μοντέλο από το Ηνωμένο Βασίλειο επενδυτικά ομόλογα κοινωνικά. Και τώρα λέμε ότι θα δαπανίσουμε τα χρήματα μόνο όταν επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Αυτό έχει άμεση σχέση με το InvestEU και τα 40 δις, ε, τα οποία για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε στο επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4 δις, όχι 40 συγγνώμη, για ε, τα κοινωνικά ζητήματα. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να συντονίσετε τα όσα θα γίνουν με το InvestEU και ε, ε, το θέμα είναι το ESF συν θα εστιάσει σε αυτή την προς, πιο πρόσφατη γενιά παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικών ομολόγων. Και μια τελευταία ερώτηση πρέπει να αντιληφθούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ είναι και μια πολύ σοβαρή πολιτική δήλωση για το τι επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντήθηκαν με την μειονότητα των Ρωμά και μας είπαν ότι πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ορισμένες φορές έχουν την αίσθηση ότι η Ευρώπη ε, δεν τους ε, λαμβάνει υπόψη. Ε, δεν τίθεται θέμα χρημάτων μόνο το γεγονός είναι ότι αυτό είναι συμβολική σημασία για μας. Πρέπει να πιστέψουμε ότι τα κοινωνικά μέσα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι επένδυση σε μια καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζάντερς τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς, ε, κυρία Σαντέρ, να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ντέβιτ Κάζα και τους κοιόδης εισηγητές για την δέσμευσή του για το θέμα αυτό. Να έρθω στο θέμα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και βρίσκονται σε επισφαλή θέση είναι θέμα το οποίο είναι πανευρωπαϊκό. Ε, ξεκινάει και το κρύο σχεδόν παντού στην Ευρώπη και θα ήθελα να σταθώ σε ένα, ένα πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους ε, περισσότερο στερημένους και να πω ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρώπη έχουμε στόχο να υποστηρίξουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει όμως καταρχάς να τα απλοποιήσουμε, να μπορούν ε, να έχουν πρόσβαση οι δικαιούχοι με πολύ πιο εύκολο τρόπο, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τις ε, πιο μικρές δομές να έχουν πρόσβαση. Και ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι ως προς το επίπεδο. Ε, πριν από κάποιες εβδομάδες είδα όλες τις ε, τράπεζες τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από τη Γαλλία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη στο Στρασβούργο και μου ανέφεραν τις ανησυχίες τους ε, για τη μείωση της χρηματοδότησης για αυτούς τους οργανώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να υποστηρίξω να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το όριο στο 3% που έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους πλέον ευάλωτους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μάντερς. Ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Σούκοβα για την παρουσίαση. Σημαντικότατο το έργο που γίνεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Μιλάμε για κοινωνικό αποκλεισμό και κυρίως τους νέους, τους άνεργους νέους. Εστιαζόμεθα σε αυτούς περισσότερο. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να πείσουμε την κοινωνία ότι είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγεται ο κοινωνικός αποκλεισμός και να υπάρχει μια ισορροπία στην κοινωνία. Τώρα, μια ερώτηση. Μπα χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μόνο για να πείσουμε τι ευρωπαϊκέ κοινωνίε ότι πρέπει να αποφευθεί ο κοινωνικό αποκλεισμό διαφορετικά. Στο τέλο, επικρατεί μια ανισορροπία σε μια ε, κοινωνία που γίνεται δυσλειτουργική. Τα τελευταία 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εσωτερική αγορά εστιάστηκε κυρίω επί πολυεθνικών και είχαν τεράστια πλεονεκτήματα. Αλλά οι εργαζόμενοι, οι εργάτε ε, δεν είδαν τα ωφέλη από μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Να βρούμε τρόπο, θα έλεγα, να πείσουμε την κοινωνία, ούτω ώστε να αποφεύγει το κοινωνικό αποκλεισμό. Εκπροσωπώ ε, το κόμμα των δικαιωμένων. Αν έχεις, αν είσαι πάνω από 50 και έχεις χάσει τη δουλειά σου, δύσκολα ξαναβρει δουλειά, είσαι πολύ ακριβώ κλπ. κλπ. Είχαμε μια ιδέα που προέρχεται από την ιστορία. Κατά το παρελθόν είχαμε τις διάφορες ενώσεις των ειδικών συντεχνίες ε, που είχαν συνδύαζαν την εμπειρία και σύγχρονη παιδεία αν μπορούμε να συνδυάσουμε λοιπόν τους νέους να βρουν δουλειά μαζί με τους πλέον ηλικιωμένους που έχουν μεγάλη εμπειρία τότε μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Και αυτή είναι μια κοινωνική ένταξη, συμπερίληψη. Αν δεν σεβαστείς τους νέους δεν έχεις μέλλον. Αλλά αν δεν σεβαστείς και τους πιο ηλικιωμένους, δεν έχεις μέλλον και πάλι. Άρα χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη κοινωνία. Αυτές λοιπόν η διπλή προσέγγιση υπάρχει. Είναι μια καλή ιδέα πώς μπορούμε να πείσουμε τις κοινωνίες μας να κινηθούν ούτως ώστε να αποφεύγεται το κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σατούρη τελευταίος. Και μετά να απαντήσει η κυρία Σούκοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Σούκοβα. Ευχαριστούμε το, το, για την παρουσίασή του. Είναι ένα εργαλείο, το Κοινωνικό Ταμείο Πλής, ούτω ώστε να έχουμε μια Ευρώπη που προστατεύει και υποστηρίζει τους πλέον αδύναμους σε μια στιγμή όπου ακόμα και το ευρωπαϊκό εγχείρημα και αυτό που αντιπροσωπεύει στους πολίτες μας να είναι καλύτερη εικόνα. Θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο ύψος των περιστάσεων τα μέσα και το, ο μηχανισμός να είναι προσβάσιμος. Επανειλημμένα έθεσαν ένα θέμα και ερώτημα οι συνάδελφοι. Τι δεσμεύσει αναλαμβάνετε για να κοινοποιήσετε ε, αυτό το ταμείο, ούτω ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των διαφορομένων, να μειωθεί τελικά η γραφειοκρατία. Ε, ε, υπάρχει καλύτερη κινητοποίηση λοιπόν των πόρων και του ταμείου. Κάποιοι φορεί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσει που υπάρχουν σήμερα, αν δεν υπάρχει απλούστευση. Τα εργαλεία είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Μόνο του μεγαλύτερου φορεί ευνοούν. Και ξέρουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, πω η σχετικότητα τη δράση τη κοινωνική είναι καλύτερη όταν είναι κοντά στα πιο χαμηλά επίπεδα. Και θέλουμε να έχουμε φορεί που είναι πιο κοντά στον απλό άνθρωπο. Ερώτηση. Ποια δέσμευση αναλαμβάνεται ώστε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί να μπορούμε να το ακοπηθούμε στις ε, ε, κατεπίγουσες ανάγκες χωρίς να υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία που δίνει και μια κακή εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά έχουμε τα μέσα. Αναφερθήκαμε στη βοήθεια για του πλέον αδύναμου, Μιλήσατε το 2%. Το Κοινοβούλιο είχε καταφέρει να πετύχει συνένεση που ήταν περισσότερο ε, στο 3% που ήταν και κόκκινη γραμμή. Υπάρχει μια ανησυχία που επικρατεί σε κάποιους οργανισμούς. Εγώ μιλάω για, το, για τη Γαλλία υποστήριξη. Λοιπόν, ανησυχούν διάφοροι φορεί. Ο, ο ίδιο ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο κ. Σασόλη, εξέφρασε ανησυχία, άκουσε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Ε, υπάρχει μείωση των πόρων γενικά και διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Σασόλη στους διάφορους φορείς ότι κάτι πρέπει να γίνει. Μπορούμε εμείς, τώρα που ξεκινάει ο τρίλογος, να διαβιβάσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στις κοινωνικές και το κατά πόσο η δυνατότητα πρέπει να είναι στο ύψος αυτό. Όταν υπάρχει επιτακτική ανάγκη, ούτως ώστε να αποδείξουμε ότι εισακούμε τους πλέον αδύναμους και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και παρεμβάσεις σας. Κυρία Σούκοβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ενεργό συμμετοχή σας, τις ερωτήσεις και απαντήσεις και τα σχόλια. Υποστηρίζετε την εντολή για διαπραγματεύσεις. Εγώ είμαι έτοιμη να ξεκινήσω τον τριμερή διάλογο. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εμπλακεί στι συζητήσει. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επιταχύνουμε τη διαργασία και να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν ο τριμερή διάλογο, να συνοψίσω τι ερωτήσει. Κάποιες από αυτές ε, συμπλήρουν μία την άλλη για τον προπολογισμό και τις διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις του πολιτές δημοσιοπικό πλαίσιο είναι δυσχερέστατες. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Δεν είμαι αισιόδοξο άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσες συζητήσεις έχουν διεξαχθεί για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν περάσει διάφορες προθεσμίες για την υιοθέτηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε τα ποσά που θα διατεθούν για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσης για την επόμενη περίοδο, αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν πρέπει να μας σταματήσει από το να συζητήσουμε τις διατάξεις, τους κανόνες και τα θέματα που δεν σχετίζονται με τα οικονομικά του κανονισμού για να προχωρήσουμε και να μην καθυστερούμε στις ε, λόγω των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το διαπραγματευτικό αυτό πλαίσιο είναι πολύ ευρύ, καλύπτει όλα τα ευαίσθητα στοιχεία για τα κράτη-μέλη και γι' αυτό οι αγγείλες και οι παρενθέσεις βγαίνουν πολύ αργούς ρυθμούς. Πολύ λίγες παρενθέσεις έχουν βγει από το κείμενο οι απαιτήσει για θεματική συγκέντρωση θα παραμείνουν ε, μέχρι τέλους, φοβάμαι. Αναφερθήκατε στο διοικητικό άχθο και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το διοικητικό άχθο. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ και η εφαρμογή της κοινή διαχείρισης ε, βαρύνει πολύ ε, τα κράτη-μέλη με ευθύνε. Τα κράτη-μέλη αναπτύσσουν εθνικούς κανόνες βάσει των οριζοντίων γενικών διατάξεων και καμιά φορά αυτοί οι κανόνες ε, είναι συμπληρωματικοί, ε, ε, δεν χρειάζονται πάντα, αλλά παρέχουν κάποια ασφάλεια και διαβεβαιώσεις για τις αρχές. Από, εφόσον συμμετέχει στη συνεδρίαση της Εποπτικής Επιτροπής κάθε προγράμματος Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάντα θέλουμε να πούμε ότι κάποιες διαδικασίε μπορούν να πλουστευτούν. Μπορώ να σας δώσω διάφορα παραδείγματα που έχω αντιμετωπίσει ίδια, όπου τα κράτη-μέλη περιπλέκουν τόσο τους κανόνες ότι είναι θαύμα που καταφέρουν να κάνουν οτιδήποτε. Νομίζω ότι καλοί την πίστη προσπαθούν να αποφύγουν κατάχρηση των πόρων και του προπολογισμού τους δεν το πετυχαίνουν πάντα αυτό, διότι τελικά εμποδίζουν πλήρω την ε, υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι συνάδελφοί μου, λοιπόν, όταν πηγαίνουν σε συνεδριάσει τη Εποπτική Επιτροπή, όταν συζητούν του κανόνε για τι επιχειρήσει και του κανόνε για υλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων, πάντα προσπαθούν να τονίσουν το πόσο θα μπορούσαν να αποφύγουν τι επίπλοκε διατάξει, να μην εμποδίζονται οι μικροί φορεί να έχουν πρόσβαση στου πόρου. Στον οριζόντιο κανονισμό έχουμε μια διάταξη σύμφωνα με τον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρώνονται εντό 60 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως για πληρωμή και την τελευταία προγραμματική περίοδο τα κράτη-μέλη το επέκτηναν στα 90, στις 90 μέρες. Οι συνομοθέτες το αποφάσισαν αυτό. Προσπαθούμε καλή και πάλι να έχουμε συντομότερη περίοδο, διότι είναι πολύ σημαντικό για τους μικρούς δικαιούχους να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση έγκαιρα. Ε, πάντα υπάρχει δυνατότητα οι επιχειρήσει να σχεδιαστούν με ένα τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε οι εφαρμοστικοί φορεί, οι εκτελεστικοί φορεί, οι δικαιούχοι και διάφοροι φορεί να παραλαμβάνουν κάποια προκαταβολή. Αλλά αυτό σχετίζεται με άλλε διατάξει για οικονομική σταθερότητα κλπ. Προσπαθούμε να πλουστεύσουμε επίση την ε, υλοποίηση των προγραμμάτων ε, του ESF-SYN με απλουστευμένες επιλογές κόστους. Αλλά είναι κάτι που τίθεται όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας στέλνει τα τιμολόγια για τις πληρωμές, αλλά ε, εάν είναι πολύ κοντά το ποσό στην πραγματική δαπάνη, μπορούν να επιστραφούν και κάποια χρήματα στους δικαιούχους, να αποζημιωθούν και δικαιούχοι. Υποστηρίζω τις προσπάθειες. Για να συνεχίσουμε την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και βλέπουμε ότι υπάρχει ουσιαστική μείωση των επιπέδων της ανεργίας των νέων. Είμαστε στο 12,9% κατά μέσο όρο πλέον. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι το 2018 το επίπεδο της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα ήταν 19,5%, λιγότερο από το 20% δηλαδή, και το υψηλότερο ποσοστό είναι στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα. Αλλά γνωρίζουμε ότι οι προσπάθειες και η πρωτοβουλία για την απασχόληση της νεολαίας ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός που ε, άλλαξε τα πράγματα. Σε πολλές χώρες η εφαρμογή και η χρηματοοικονομική στήριξη οδήγησε σε πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές ε, για τον τρόπο που παρέχονται οι υπηρεσίες στους νέους. Χρειάστηκε χρόνος όμως για να γίνει κατάλληλη προσαρμογή και να το παρέχουμε στους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι προσπαθούμε να προσελκύσουμε τους περισσότερο αδρανείς νέους ανθρώπους και αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, θα είναι δύσκολο και θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή ε, των εταίρων, μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των οργανώσεων που μπορούν να καθοδηγήσουν ανθρώπους που είναι αδρανείς και δεν ενδιαφέρονται καν να βρουν μια θέση εργασίας ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή να λάβουν κάποιο πιστοποιητικό για τις δεξιότητές τους. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι με αυτό το πολύ χαμηλότερο ποσοστό ανθρώπων που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, κατάρτιση ή ε, ε σπουδές, ε, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Με τον Επίτροπο ε, μπορώ να πω ότι υπάρχουν δράσεις και πράγματα τα οποία έχουμε εξετάσει για να αναβιώσουμε τις πρωτοβουλίες αυτές και να επεκτείνουμε το εργαλείο αυτό που θα έχει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι τώρα. Νομίζω ότι για την εγγύηση για τα παιδιά που είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Δεν υπάρχει πλαίσιο πολιτικής, ε, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ε, κονδύλια για τα παιδιά και γίνονται δαπάνες βάσει των ε, συστάσεων του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2000, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030. Υπάρχει λοιπόν μια πολιτική που υποστηρίζει μια σειρά αποδράσεις για τα παιδιά στην Ευρώπη, αλλά θα αν απτυχθεί και μια εγγυηση για τα παιδια οπως ε, υποσχεθηκε η σαν προεδρος και αυτο θα βασιστει και σε ενα σκοπιμότητας ε, για να δούμε ποιες είναι οι ομάδες στόχος, ε, οι οποίε θα πρέπει να εξετάσουμε στο μέλλον, πώ θα διαπιστώσουμε ποιε είναι οι ομάδε αυτές, τι είναι το πλέον κατάλληλο για αυτούς, ώστε ε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αναπτύξουμε το πλαίσιο. Ε, όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική ένταξη με διάφορα μέτρα και μέσω των ε, συγκεκριμένων στόχων που έχουμε και των 11 στόχων και εξετάζουμε πώς λαμβάνονται υπόψη τα άτομα με αναπηρία για όλους τους συγκεκριμένου στόχους, ε, είτε για ε, δράση για την απασχόληση, πρόσβαση στην εκπαίδευση ή κοινωνική ένταξη. Και θεωρώ ότι τα μέτρα για την κοινωνική ένταξη μπορεί να ε, τα μέτρα για την απασχόληση μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνική ένταξη όταν αποκτήσει κάποιος τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες. Κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν και στο ταμείο για τους ε, πιο ευάλωτος. Να σας πω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είναι ένα μικρό ταμείο, αλλά προσπαθούσαμε να έχουμε μια πολύ απλή προσέγγιση, να είναι πολύ εύκολη πρόσβαση και να είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του κάθε κράτους μέλος. Ε, αφήσαμε πάρα πολλές ανοιχτές δυνατότητες, ώστε το κάθε κράτος μέλος να επιλέξει ποια θα είναι η ομάδα στόχος, τι είδου στήριξη θα παρέχει, ε, πόσο συχνά θα παρέχετε στήριξη, με ποιες ε, οργανώσεις ε, τέρους, ενδιάμεσους φορείς. Ήταν ένα πάρα πολύ ευέλικτο μέσο και πρέπει να πω ότι σε κάποιες χώρες ήταν πραγματική επιτυχία. Βλέπουμε τα κράτη-μέλη που ε, είχαν ελάχιστα ποσά ε, στην αρχή, ε, εξετάζουν πολύ ψηλές αυξήσει διότι είδαν ότι υπάρχει πραγματικά προστιθέμενη αξία και έγινε και μια ενδιάμεση αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε προ τα τέλη του προηγούμενου έτου και δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό αυτή τη στιγμή καλύπτει και μια υποχρέωση ε, από όσου παρέχουν ηλική στήριξη να ε, υπάρχουν και συνοδευτικά μέτρα. Στο μέλλον, επειδή θα συμπεριληφθεί στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ, θα χρησιμοποιήσει τι παραδοσιακές προτεραιότητε επενδύσεων για αυτή τη μορφή στα συμπληρωματικά μέτρων. Οτιδήποτε λοιπόν προβλέπεται για ηλική υποστήριξη βάση του στόχου 11 είναι για υλική στήριξη. Δεν θα δίνεται για συνοδευτικά μέτρα, συμπληρωματικά ή οτιδήποτε άλλο. Και θα είναι και ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος να προσεγγίσουμε ε, όλους ε, όσοι είναι αποκλεισμένοι και θα είναι και ένα πρώτο βήμα να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία ή να τους βοηθήσουμε αν έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να ε, επιστρέψουν στην εργασία. Θεωρώ λοιπόν ότι οι οργανώσεις των τραπέζων τροφίμων δεν θα πρέπει να ανησυχούν διότι δεν υπάρχει ουσιαστική μείωση και θα είναι πάνω από το 4% που είναι ο στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνολικά. Και νομίζω ότι ένα από τα επιπλέον ε, στοιχεία του Ταμείου για τους πιο στερημένους είναι ότι μπορέσουμε να στηρίξουμε και να χρησιμοποιήσουμε οργανώσεις εταίρους ε, ε, ως ενδιαμέσους για να προσεγγίσουν ε, τους ανθρώπους αυτούς. Αυξήσαμε τις δυνατότητές τους, την εμπιστοσύνη τους, αλλά και την εμπιστοσύνη και πιθανών δωρητών. Και υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες λαμβάνουν και ε, χορηγίες, δωρεές, οι οποίες χρησιμοποιούν αυτές τις οργανώσεις ως διάβλο για να φτάσουν τα χρήματα αυτά στους φτωχούς ανθρώπους. Σε κάποια κράτη-μέλη, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου δεν υπάρχουν τράπεζες ε, τροφίμων, οδήγησαν στην ε, δημιουργία τραπεζών τροφίμων. Είναι λοιπόν ένα επιπλέον ε, πλεονέκτημα αυτό. Βέβαια, οι τράπεζες τροφίμων πρέπει να ρυθμιστούν σε κάποια κράτη-μέλη. Πέρασε νομοθεσία για πρώτη φορά επί του θέματος και νομίζω ότι η άμεση βοήθεια, η ηλική συνδρομή που δίνει στα παιδιά θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο με την ηλική υποστήριξη, αλλά και μέσω αυτών των οργανώσεων και των ενδιαφερομένων και ενίσχυσή τους. Όταν ε, θεωρούμε ότι δεν γίνεται σωστή η χρήση πόρων, τότε παρεμβαίνουμε. Κάνουμε τους ελέγχους μας, ε, σταματάμε πληρωμές, κάνουμε χρηματοπιστωτικές αλλαγές, ανάλογα με το είδος των παρατεπιών, έχουμε μορφές παρέμβασης διάφορες. Νομίζω ότι είναι πολύ αποτελεσματικό το σύστημα ελέγχου μας και έχει υπάρξει μεγάλη βελτίωση στην λειτουργία των αρχών ελέγχου. Γι' αυτό στον κανονισμό για τις κοινέ προβλέψεις λέμε ότι όταν υπάρχει, όταν, όπου υπάρχει μια αξιόπιστη αρχή ελέγχων, τότε παρεμβαίνει λιγότερο η Κομισιόν. Τώρα για τις ε, κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική απασχόληση. Σε κάποια κράτη-μέλη έχουν γίνει περισσότερα και ξέρουν πολύ καλά πώ να δημιουργήσουν αυτέ τι κοινωνικέ επιχειρήσει, πώ να την βοηθήσουν να λειτουργήσει. Ενώ σε άλλα κράτη-μέλη δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει διεθνική συνεργασία. Για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, για εννέα θέματα συζητάμε κοινέ προκλήσει που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Και Έχουμε πολύ καλά παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων και τέτοιων μορφών απασχόλησης. Μπορούμε να σας στείλουμε ένα συμπίλημα για το πόσο έχουμε βοηθήσει στα θέματα αυτά να ξεκινήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις και να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν. Συμφωνώ ότι η υποβολή εκθέσεων, η επιτήρηση και η παρακολούθηση είναι πολύ καλή μέθοδος. Έχουμε δείκτες και για ενδιάμεσες φάσεις και για το τελικό αποτέλεσμα για να μετρήσουμε όχι μόνο την άμεση επίπτωση οποιασδήποτε παρέμβαση, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα μετά από 6 και 12 μήνες. Ρωτήσατε για τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Από τα 2,5 δισεκατομμύρια Το 1,1 αφορούσε την ε, μακροχρόνια ανεργία, αλλά θα πρέπει να ελέγξω, δεν είμαι σίγουρη. Αναφέρθηκα στην επιτήρηση στην οποία συμμετέχουμε και ορισμένε φορέ παρεμβαίνουμε για την αξιολόγηση. Είναι μόνο ex post. Τα κράτη-μέλη δεν ήθελαν ε, ενδιάμεσες. Αλλά το σύστημα υποβολής εκθέσεων θα αλλάξει στο μέλλον. Δεν θα υπάρχουν αιτήσει εκθέσει εφαρμογή που γίνονται λοιπόν μια φορά το χρόνο. Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν εκθέσει με πιο διαρθρωμένο τρόπο κάθε δύο μήνε για το τι πρόοδο έχει επιτευχθεί όσον αφορά και τα υλικά αποτελέσματα και τη χρήση των πόρων. Έτσι θα έχουμε στοιχεία πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα, πολύ πιο ε, έγκαιρα. Διότι οι δείκτες μας για την ε, κοινή ε, αποτελεσματικότητα καλύπτουν την ηλικία, το χρόνο ανεργίας, ε, το φύλλο. Πιστεύουμε ότι βοηθάμε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα φύλου. Η έξποστα αξιολόγηση ε, απέδειξε ότι οι παρεμβάσεις μας, ε, οι παρεμβάσεις δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πηγαίνουν κατά 5% στους άνδρες και 50% στις γυναίκες. Ε, με την Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΗΝ εργαζόμαστε για να προχωρήσει το κοινωνικό παράθυρο για τις κοινωνικές επενδύσεις και τις δεξιότητες στα πλαίσια του InvestEU. Και εργαζόμαστε και για τις καθεντήρες γραμμές που θα είναι τμήμα των οδηγιών, για τους κανόνες, για το παράθυρο κοινωνικών επενδύσεων του InvestEU πάντα. Έχουμε πολλές δυνατότητες. Ένα τεράστιο αριθμό δυνατοτήτων για να συμπληρώσουμε τη δράση του ESF-SYN όπου χρειάζονται για παράδειγμα υποδομές για κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες. Για την ενεργό γύρανση. Ε, όλοι μεγαλώνουμε, έχουμε πολλές γνώσεις και δύναμη λόγω της εργασίας. Σε κάποιες ε, βόρειες χώρες έχουμε πραγματικά πολύ καλά παραδείγματα. Ηλικιωμένοι μετά από κάποια ηλικία, ανάλογα βέβαια και με την υγεία τους, εργάζονται μαζί με νέους. Έχει γίνει σε κάποια κράτη-μέλη, είναι απόλυτα δωρεάν. Πολλά μέτρα μπορούμε να ε, στηρίξουμε μέσω του esf sin Εξαρτάται από το κράτος μέλος. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, τι, στόχους θέλει τι μέτρα θέλει να εφαρμόσει. Αλλά η πείρα που έχει ένα άτομο που έχει εργαστεί 30 χρόνια είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη. Και δεν αρκεί απλώς ε, να αφήσει ένα σημείωμα από την πύρα του. Πρέπει να βοηθήσουν οι ηλικιωμένοι για να βοηθήσουν ε, τους νέους που έχουν κάποια κατάρτιση αλλά δεν έχουν πείρα να ενταχθούν στον κόσμο της εργασίας. Φυσικά, τέτοια προγράμματα κοινή απασχόληση νέων και ηλικιωμένων που συμβαίνει ήδη σε κάποια κράτη-μέλη, όχι παντού, βοηθάνε πολύ. Αλλά βέβαια είναι δύσκολη η εισαγωγή του. Δεν τα εισάγουμε εμεί. Έχουμε περιορισμένε εξουσίε ε, έναντι των κρατών μελών. Απλώ να... επιχειρούμε να βοηθήσουμε μέσω απλούστευση και των διαδικασιών. Αλλά πρέπει να σα πω ότι ασχολούμαι εδώ και 8 χρόνια με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχει αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων και το σύνθημά μας ότι δεν αφήνουμε κανένα στο περιθώριο θα εξακολουθήσει να ισχύει. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα πιο ευάλωτα άτομα φυσικά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει και το εργατικό, το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται η οικονομία μας και οι δεξιότητες που χρειάζεται η οικονομία μας, ούτω ώστε όλοι να εργαστούμε για μια καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας σήμερα. Πραγματικά σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων Ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα κυρία Σούκοβα. Η ερώτησή μου προς τον κύριο Κάζα. Αν θέλει να του δώσω το λόγο για να κάνετε ένα κλείσιμο. Παρακαλώ. Όχι. Ωραία. Καλώς. Ευχαριστώ και από πλευράς μου λοιπόν. Νομίζω ότι κατέστη σαφές ε, τι σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για ε, μεγάλο χρονικό διάστημα ήμουν τοπικά εκλεγμένη και κάθε φορά που υπήρχαν προβλήματα οι δήμοι και οι κοινότητες ε, είχαν πρόβλημα για να λάβουν πρωτοβουλίες. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Οπότε κλείνουμε το θέμα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, οπότε τελειώνουμε. Από πλευράς μου δεν έχω καμία περαιτέρω ανακοίνωση. Απλώς να σας πω ότι η επόμενη συνεδρία θα γίνει 14 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και σας εύχομαι καλό βράδυ. Και σε εσάς κυρία